η υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν βάσει τη συνήθω νομοθετική διαδικασία, να σα ενημερώσω ότι μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, ο πρόεδρο την Δετάτη θα υπογράψει εννέα πράξει, οι οποίε εγκρίθηκαν βάσει τη συνήθω νομοθετική διαδικασία, βάσει του άρθρου 78 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι των πράξεων αυτών θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση.